μερίσες διάταξης ε, είναι η έκθεση της κυρίας Λίδια Γκέριγκερ Ντεόντεμπερκ με θέμα την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροδιαφορών και τη διαδικασία έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής. Παρακαλώ την εισηγήτριά μας, την κυρία Γκέριγκερ Ντεόντεμπερκ. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Με την αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για αποτελεσματικότερους και ταχύτερους μηχανισμούς ε, επίλυσης των μικροδιαφορών μεταξύ μεμονωμένων ε, πελατών είτε και μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να τονώσουμε την ε, οικονομική ανάπτυξη. Η διαδικασία αυτή, η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών προβλέπει αύξηση του, του κατωτάτου ορίου από 2.000 σε 10.000 ευρώ και στόχο έχει την απλούστευση κυρίως της διαδικασίας ε, διασυνοριακών μικροδιαφορών εμπορικού και οικονομικού χαρακτήρα και επίσης συντομεύει την ε, προθεσμία εκδίκασης από 2 χρόνια και 5 μήνες σε 5 μήνες και μειώνει το κόστος των μικροδιαφορών κατά 40%. Μάλιστα, η με τη διαδικασία αυτή και με την αύξηση του ορίου αυξάνει και τον αριθμό των ε, μεμονωμένων προσώπων αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μπορούν να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους. Ε, χαίρομαι γιατί μετά από 1,5 χρόνο συζήτησης ε, με το Συμβούλιο καταλήξαμε στέναν κανονισμό που τώρα στη διάρκεια της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας ορίμασε και κατέληξε στη φάση της ψηφοφορίας. Πιστεύω ότι η νέα ευρωπαϊκή διαδικασία επίλυσης μικρών διαφορών θα βοηθήσει τους πολίτες ώστε πιο αποτελεσματικά, πιο γρήγορα και πιο φθηνά να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους. Γιατί έχουμε δισεκατομμύρια αξιώσεις μικρών όμως ποσών και μάλιστα οι πολίτες δεν είναι γυρουναγωγές γιατί είναι αποτρεπτικό το κόστος για την εκδίκαση τέτοιων αποφάσεων. Έτσι, οι πολλές επιχειρήσεις ε, ατιμόρυτα μπορούν να εξαπατούν τους, τους ε, πελάτες τους. Επίσης, με την απλούστευση των διαδικασιών, χωρίς ε, περιττή μετακίνηση σε τρίτη χώρα και χωρίς πρόσληψη δικηγόρου στην άλλη χώρα, μπορούμε μέσω εφαρμογής εικονοδιασκέψεων, τηλεδιασκέψεων ή εξαποστάσεως επικοινωνίας να μειώσουμε το κόστος αυτής της εκδίκασης. Επίσης γίνεται δυνατότητα πληρωμής ε, με χρεωστική ή πιστοτική κάρτα. Δεν απαιτείται μετάφραση σε όλες τις γλώσσες. Αρκεί ένα πιστό αντίγραφο της απόφασης και ε, μία σύντομη μετάφραση ενός τμήματος μόνο της βεβαίως Έτσι μειώνεται το κόστος ε, που δεν είναι πια δυσανάλογο σε σχέση με το ύψος της αξίωσης, το ποσό της αξίωσης. Ήταν πολύ θετική η συμφωνία με το Συμβούλιο και καλύπτει κάποια στοιχεία και του εργασιακού δικαίου και ενισχύει και την ε, καλύτερη διακίνηση των ε, εργαζομένων. Δυστυχώς έμεινε ανέδοτο το Συμβούλιο σε αυτό και παρόλα αυτά έχουμε μια ρήτρα ε, και για την αύξηση του ορίου των αξιώσεων αλλά και για, το, για την περίοδο της εκδίκασης. Με βάση τη νέα απλουστευμένη διαδικασία που θα ε, τεθεί σε εφαρμογή ε, έξι μήνες μετά την θέση ισχύ του κανονισμού, ε, πολλές αξιώσεις θα ικανοποιηθούν και ελπίζω έτσι να σταματήσουν οι μαζικές εξαπατήσεις των πελατών από επιχειρήσεις. Ευχαριστώ θερμότατα όλους τους κοιόδης ηγητές για την αγαστή συνεργασία που είχαμε, την, τους εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, τους βοηθούς μου ε, και τη γραμματεία της Νομικής Επιτροπής. Πιστεύω ότι με τον νέο κανονισμό ε, θα έχουμε πολύ καλύτερη βελτίωση. Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπούντα, τους, τους προηγούμενες προεδρίες, την Λετωνική, και τους αρμοδίους ε, υπουργούς που συνέβαλαν στην ε, διεκπαιρέωση αυτού του θέματος. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους βοηθούς μου, Μόρτοβαν, Τζαρβόνιες και Κις. Σας ευχαριστούμε, κυρία Γκέριγκερ. Και ευχαριστώ θερμά που τηρήσατε και το χρόνο σας, παρά το περίπλοκο του θέματος. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην ε, Επίτροπο Γιώροβα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κάθε μέρα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις συνάπτουν για συνοριακές ε, πράξεις. Και βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την εμπορική δυνατότητα οι Ευρωπαίοι πολίτες όταν δεν τους παραδίδονται αυτά τα οποία έχουν παραγγείλει ή είναι λατωματικά τα προϊόντα αυτά. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και να ε, εκφράσουν και να επιβάλλουν τα δικαιώματά τους. Έτσι λοιπόν προσφέρουμε μια ενιαία δυνατότητα να γίνεται αυτό με φθηνότερο και πιο ταχύ τρόπο. Το τρέχον σύστημα λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια. Εμείς το αξιολογήσαμε και έχουμε εντοπίσει ποιες ελλείψεις έχει και τώρα έφτασε η ώρα για να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την κυρία εισηγήτρια όπως επίσης και όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την συνεργασία που είχαμε στο θέμα αυτό. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό τόσο γρήγορα μάλιστα. Ο στόχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να εξυγχρονίσουμε αυτή τη διαδικασία επίλυση μικροδιαφορών, να επεκτείνουμε την εφαρμογή τους μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ. Και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη όσον αφορά final compromise sets the threshold 5,000 Currently, it is only 2,000 Για τις ε, περιπτώσεις των 2.000 ευρώ αυτών των μικροδιαφορών. Γνωρίζω ότι κάποιοι από εσάς βεβαίως θα θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν αυτές οι διαφορές από μέρους των εργοδοτών να είχαν συμπεριληφθεί. Θα επανέλθουμε όμως στο μέλλον σε αυτήν την ε, κατηγορία διαφορών αφού εξετάσουμε και όλες τις υπόλοιπες πτυχές της. Σκοπός μας είναι να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση, πιο αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Βεβαίως, έχουν καθοριστεί τα πλαίσια και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποθαρρύνονται οι πολίτες από το να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Και αυτό βεβαίως συμπεριλαμβάνει και τις περιπτώσεις των διακανονισμών, των συμβιβασμών και πάντα προς όφελος της προάσπισης των συμφερόντων των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Η ο αναθεωρημένος ε, κανονισμός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνοδεύεται από μία ενημερωτική καμπάνια και από τη διάδοση όλων των αντίστοιχων πληροφοριών. Σα ευχαριστώ. Uh, on behalf, uh... Και τώρα οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Πρώτα εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ο κύριος Μπούτα. Δύο λεπτά. Domnule președinte, doamna comisar, doamnelor și domnilor colegi. Îi mulțumesc. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή για την, την εισηγητρία για την μεγάλη συνεργασία και για και την Επιτροπή αλλά και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή την έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη χρειάζεται λοιπόν ε, έναν ιερό χώρο στην Ευρώπη και απλοποιημένε διαδικασίε. Οι Ευρωπαίοι πολίτε θα επωφεληθούν σημαντικά από αυτέ τι απλοποιημένε διαδικασίε σε ό,τι αφορά την επίλυση μικροδιαφορών έω 5.000 ευρώ. Δεν θα υπάρχουν εθνικά σύνορα για τα για τους ιδιώτες αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και πληρωμών θα καταστούν αποτελεσματικά εργαλεία και ο ορισμός των διασυνοριακών υποθέσεων θα διευρυνθεί και θα περιλάβει και περαιτέρω στοιχεία. Τα τέλη και οι φόροι θα πρέπει να είναι αντίστοιχα της αξίας της συναλλαγής για να μην είναι απαγορευτικά για τους πολίτες και η καλή πίστη στις ε, εμπορικές συναλλαγές θα βελτιωθούν. Η νομική βεβαιότητα και η νομική ασφάλεια θα ενισχυθεί επίσης. Με την πρωτοβουλία λοιπόν αυτή θα δημιουργηθούν ίσοι όροι για όλους. Σε όλο τον ενιαίο αυτονομικό χώρο τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να εφαρμόσουν τον κανονισμό αυτό και σε επίπεδο εθνικών κρατών θα δημιουργηθεί αυτή η πραγματικότητα Πολύ λυπάμαι που δεν μπορέσαμε να διευρύνουμε τον κανονισμό αυτό προκειμένου να περιλαμβάνει και την νομοθεσία για την, ε, τα εργασιακά. Προκειμένου και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα απλοποιημένα μέσα για να ανακτούν οι εργαζόμενοι. Δηλαδή τα χρήματα από τους εργοδότες μπορούν να τον επιβεβαιώσουν. Αυτό θα ενισχύσει και τη φοροδιαφυγή και τη μαύρη εργασία. Αλλά είμαι πεπισμένο ότι στο μέλλον όλα τα ευρωπαϊκά τεχνικά όργανα θα βρουν μια λύση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πρόεδρο. Εξ ονόματο τώρα του ECR, ο κύριο Τζαμπάσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Γκέριγκερ για την έκθεση και για τους συμβιβασμούς. Η πολιτική μας ομάδα υποστήριξε τους συμβιβασμούς στην Επιτροπή. Το 2012 Υιοθετήθηκε εμπλουστευμένη διαδικασία. Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, η Κομισιόν θα πρέπει να παρουσιάσει μια λεπτομερή έκθεση για το πώς λειτουργεί η διαδικασία αυτή. Αυτή η αναθεώρηση είχε ως στόχο να καταστήσει αυτή τη διαδικασία πιο ελκυστική στους Ευρωπαίους πολίτες. Πιστεύω ότι με κοινέ προσπάθειες μπορούμε να πετύχουμε αυτό τον κοινό στόχο. Το αυξανόμενο κατόφλι από τα 2.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ είναι επίσης κάτι πρόσδεκτο. Θα βοηθήσει τους πολίτες και τις μικρές και μέσες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ομάδας Άλντε, ο κύριος Μαρίνιο Πίντο. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εξ ονόματος της ομάδας μου να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έργο της και να υπενθυμίσω ότι η πρωτοβουλία επικαιροποίηση αυτού του κανονισμού ανήκει στη δική μου πολιτική ομάδα, τους φιλελευθέρους, το 2011 μέσω της κυρίας Διάνας Γόλης ο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που δεσπίζει μια ευρωπαϊκή διαδικασία ε, για τις μικροδιαφορές μικρών ποσών θέλει ως στόχο να επιταχύνει ε, τις αγωγές για τα μικρά ποσά σε διασυνορικές υποθέσεις. Και συγκεκριμένο στόχος είναι να βοηθηθούν οι καταναλωτές και μικρές και μισές επιχειρήσεις εγγυόμενο την πρόσβαση στη δικαιοσύνη με ένα ταχύτερο και εύκολο τρόπο. Αυτός ο στόχος δεν μπορεί να χαθεί ε, στη γραφειοκρατία των Βρυξελών που πολλές φορές αφήνει τους πολίτες και τις μικρές επιχειρήσεις χαμένους στην πολυπλοκότητα των διαδικασιών. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι αυτό το έργο τη απλούστευσης και της προσέγγισης των πολιτών και των επιχειρήσεων στη δικαιοσύνη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο έργο που σχετίζεται με την πρωτοβουλία των φιλελευθέρων για την καλύτερη νομοθεσία. Η ευρωπαϊκή διαδικασία ε, μικροδιαφορών μπορεί να στεφτεί με επιτυχία μόνο αν το γνωρίσουν οι καταναλωτές, ε, οι επιχειρήσεις, ε, τα δικαστικά όργανα και οι φορεί παροχή συμβουλό. Τα στοιχεία που μα δίνει η Κομισιόν μας δείχνουν ότι το 85% των πολίτη και σχεδόν το ίμιση των δικαστικών οργάνων δεν ήξεραν καν ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία. Επίση πρέπει να μειώσουμε το κόστο και να αυξήσουμε την ταχύτητα τη λήψη αποφάσεω κυρίω από την πλευρά των δικαστηρίων. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ονόματος της ε, ΓΚΟΕ, ο κύριος Μάστακα, έχετε λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητούμε για τις τροπολογίες που πρέπει να υποβληθούν όσον αφορά τις σταθερές ε, και τακτικές διαδικασίες. Ο σκοπός μας εδώ είναι να βοηθήσουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλύτερη προστασία και πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ιδίως όταν πρόκειται για διασυνοριακές διαφορές. Η διαδικασία αυτή υπάρχει από το 2009 ως ε, ένα βαθμό καλυπτόταν κάποιες από αυτές τις διαφορές και υπήρχε Εξάλλου και ο αποτρεπτικός ε, χαρακτήρας αυτής της διαδικασίας. Αυτά τα 2.000 ε, ευρώ, το ανώτατο όριο αυτό που είχε τεθεί, είναι βεβαίως ε, μόνο ένα μικρό τμήμα αυτών των διαφορών. Και ο συμβιβασμός αυτός ουσιαστικά καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των υπόλοιπων διαφορών και πραγματικά διευκολύνει την πρόσβαση στην δικαιοσύνη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον εισηγητή και όλους όσους βοήθησαν για να προχωρήσει αυτή η εργασία. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος των, της EFDT, η κυρία Φεράρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφοι, πολλέ φορέ οι πολίτε και μικρέ και μισέ επιχειρήσει ε, δεν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη επειδή είναι πολύπλοκη και δαπανηρή η διασυνοριακή δικαστική διαδικασία. Ε, η Ευρωπαϊκή Διαδικασία Μικροφεφορών ε, είχε ω στόχο να πλουστεύσει και να διευρύνει περισσότερο του τρόπου πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ένα φιλόδοξο στόχο που συμμεριζόμαστε. Η πρόταση τη Κομισιόν ήταν ήδη εκτιμητέ Επιτροπή Γιούρι με μόνο εξαίρεση για τα ποσά που είχαν τεθεί ε, έχει βελτιώσει το κείμενο, βελτιώνοντας και τις δικονομικές διαδικασίες ενάντια των πολιτών. Ε, πολύ συγκεκριμένα όταν μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν τα ανάλογα οικονομικά μέσα. Όμως δυστυχώς εδώ βλέπουμε να γίνεται ένα βήμα προς τα πίσω. Δεν συμφωνούμε με το όριο των 5.000 ευρώ και ουσιαστικά υπήρχε ε, και ένας όρος όπου θα παλασσόταν κάποιος από το να πληρώσει τα τέλη του δικαστηρίου αν είχε το ελάχιστο δισόδημα. Ε, δυστυχώς ε, εδώ ε, θέλαμε να συμβάλλουμε στο να επιταχύνουμε τις διαδικασίες αυτές, αλλά δεν τα καταφέραμε. Σας ευχαριστώ, κύριος Λεμπρέτον, εξ ονόματος του ΕΝΕΦ. E Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αυτό το κείμενο ουσιαστικά βελτιώνει την κατάσταση όσον αφορά τις διαφορές κάτω των 5.000 ευρώ για συνολικές διαφορές που αφορούν κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω όμως ότι η τύχη του θα είναι η ίδια με αυτή του προηγούμενου κειμένου που κάλυπτε τις διαφορές κάτω από 2.000 ευρώ γιατί στο πνεύμα και στις συνήθειες των Ευρωπαίων η δικαιοσύνη συνεχίζει να είναι θέμα εθνικό, αρμοδιότητα εθνική. Κοιτάξτε παραδείγματος χάρη τον αριθμό των ε, δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κάτι το οποίο προσπαθεί να αλλάξει με το ζόρι, με βία προσπαθούν βάσει του άρθρου του δικαστηρίου ΤΑΦ 672, κάτι που μας δείχνει πως πραγματικά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλά και οι δικαστές είναι τελείως αποκομμένοι από την πραγματικότητα. Σήμερα βλέπουμε αυτή η φιλελεύθερη λογική η οποία συνεχίζει παρόλη την κρίση που μαστίζει την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σένφελτ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και όλους όσοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για την ε, καλή κατάληξη του, της έκθεσης για την επίλυση μικροδιαφορών. Οι τροπολογίες θα έχουν δύο συνέπειες. Καταρχάς, η διαδικασία θα είναι πιο καθολική και πιο αποτελεσματική. Κατά δεύτερον, θα καταστεί πιο ελκυστική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους ιδιώτες. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι να αυξηθεί το όριο στα 5.000 ευρώ και κατά δεύτερο επιβάλλεται υποχρέωση στα δικαστήρια να ε, χρησιμοποιούν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνίας. Έτσι λοιπόν οι τροπολογίες αυτές κρίνουν ότι θα αυξήσουν την ελκυστικότητα του μηχανισμού αυτού και θα μειώσουν και το κόστος για τους διαδικούς. Επίσης θα περιορίσουν τα, το κόστος ε, των ταξιδιών και το κόστος για τις ακροάσεις, συμμετοχή σε ακροάσεις. Τέλος, το μέσο αυτό θα μπορέσει να καταστεί με τον τρόπο αυτό πιο ευρέως ε, ε, λειτουργικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα έχει ως συνέπεια ότι θα πληρωθεί ένα χάσμα που υπήρχε στο νομικό σύστημα. Γιατί στην παρούσα φάση πολλοί επιχειρηματίε, πολλοί ιδιώτες, πολλοί απλά θεωρούν ότι δεν αξίζει τον κόπο να παρουσιαστούν, να προσφύγουν στο, στα δικαστήρια δεδομένου και του κόστους εκδίκασης. Το πιο σημαντικό λοιπόν τώρα θα ήταν να προωθήσουμε τη διαδικασία αυτή γιατί πραγματικά έχουμε καταρτήσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο το οποίο το γνωρίζει λίγος κόσμος όμως. Θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τον κόσμο να ανοίξει μικρές επιχειρήσεις γιατί ενδεχομένως να καταλαγιάσει φόβους για το κόστος προσφυγής στα δικαστήρια, ακόμα και αν πρόκειται για μικροποσά τα οποία διεκδικούν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προωθήσουμε το εργαλείο αυτό μέσω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και του κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λεκή Πρόεδρος. Επόμενος είναι ο κύριο Κοφεράτη. Για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αυτός ο κανονισμός αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη διάθεση των πολιτών και των μικρών και μέσων επιχειρήσεων και εδώ έχει βρεθεί μια συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και είναι κατηθετικό γιατί διευρύνουν το πεδίο εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του κανονισμού και μπορούν να γίνουν ίσως και καλύτερα βήματα στο μέλλον. Το σημαντικό αποτελεσμένα για το Κοινοβούλιο γιατί έχουμε βελτιώσει επί των διαδικασιών και είναι πιο αποτελεσματικό ο κανονισμό για του πολίτε και τι επιχειρήσει. Αυτέ οι διαδικασίε μπορούν να εφαρμοστούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ προσθέτουμε και τα βήματα προ τον μπρο ε, σε αυτή την πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. το χάρη σε σχέση ε, με την κατάσχεση ε, των αγαθών όσων οφείλουν. Μπορεί αυτέ οι αλλαγέ να φαίνονται ίσουν σημασίε, σημαντικέ για να δημιουργήσουν στου πολίτε στην πραγματική αντίληψη ότι αποτελούν μέρος μιας κοινότητα, μέρος ενός κοινού σχεδίου και για να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωή του, τι ηλικίε σε ένα περιβάλλον όπου οι σχέσει και οι διασυνοριακέ δραστηριότητες ε, είναι όλο και πιο συχνέ εντό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά είναι και πιο συχνέ οι δικαστικέ υποθέσει που έχουν διασυνοριακές συνέπειες. Έτσι λοιπόν τώρα χρειάζεται να εφαρμόσουμε αυτούς τους κανόνες ξεκινώντας από την απαντήση να δώσουμε έσκατες απαντήσεις στις διασυνοριακές ανάγκες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπέντ για ένα λεπτό έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμείς από το ECR έχουμε σαφές, σαφείς ε, προδιαγραφές και ε, φανταζόμαστε με συγκεκριμένο τρόπο αυτό το νομικό μέσο. Είμαστε επικριτικοί αλλά με θετική διάσταση. Θέλουμε να λειτουργεί καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά λοιπόν έχουμε να επικρίνουμε γιατί πιστεύουμε επί της αρχής ότι θα πρέπει να περιοριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί όπου έχει προστιθέμενη αξία. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε με χαρά να πούμε ότι πρόκειται πραγματικά για μια τέτοια περίπτωση. Γιατί με την προτινόμενη διαδικασία δημιουργούνται πρότυπα ε, ενοποιούνται διαδικασίες οι οποίες ιδάλλως με τις εθνικές ρυθμίσεις για τους ιδιώτες αλλά και για τις επιχειρήσεις ε, μέχρι σήμερα σήμαιναν μεγάλα προβλήματα. Ε, πρόκειται λοιπόν για έναν τομέα όπου πραγματικά δημιουργεί προστιθέμενη αξία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζουμε λοιπόν το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να άρουμε μικροδιάφορες γιατί Ω τώρα η διαδικασία αυτή υποστηρίζονταν με ηλεκτρονικό τρόπο και ελπίζουμε βέβαια οι διαδικασίε αυτέ να μπορέσουν στην πράξη να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο που προκειμένου να είναι εύκολα ε, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα και σταματάω γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να τελειώσω. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Πολύ σας ευχαριστώ που ολοκληρώσατε. Επόμενος, ο κύριος Σβόμποτα για δύο λεπτά έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, με μεγάλη χαρά είδα ότι στον τριμερή διάλογο μπορέσαμε να επεξεργαστούμε και να ολοκληρώσουμε αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους συναδέλφους από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων γιατί πραγματικά από κοινού πετύχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Θεωρώ ότι Πρόκειται για ένα τρανό παράδειγμα νομοθεσίας, το οποίο δεν είναι βεβαίως ε, πολύ ελκυστικό για το κοινό. Ε, είναι όμως σίγουρα κάτι που θα είναι χρήσιμο και θα βελτιώσει τη θετική εικόνα στους Ευρωπαίους πολίτες ε, για την νομοθεσία που παράγουμε εδώ στην Ευρώπη. Πραγματικά λοιπόν η επιτάχυνση, η απλοποίηση της διαδικασίας, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων ε, είναι εξαιρετικά σημαντικά σημεία. Την ίδια ώρα η χρήση νέων εργαλείων και μέσων για να είναι πολύ πιο αποτελεσματικές οι επιλύσεις ε, των διαφορών ιδιαίτερα σε νοριακά ε, προβλήματα βλέπουμε ότι όλες αυτές οι προσπάθειες είναι θετικές. Γιατί για κάποια κρατημέλη 10.000 ευρώ δεν θεωρείται μία μικρό διαφορά. Ακριβώς αυτές οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών είναι κάτι που σίγουρα μπορεί να μας οδηγήσει και σε κάποιες τροποποιήσεις του κειμένου στο μέλλον, ιδιαίτερα όσον αφορά την κατηγορία των διαφορών που δεν ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ και ελπίζω και στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτή την επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπόζαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι αλλαγές στην νομοθεσία είναι σημαντικές για τους καταναλωτές ε, σε μια κατάσταση όπου ένας καταναλωτής αγοράζει κάτι μέσα του διαδικτύου από μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και ανακαλύπτει ότι έχει εξαπατηθεί. τότε συνειδητοποιεί ότι το κόστος της προσφυγής στο δικαστήριο μπορεί να είναι πολύ ψηλό και στο μέλλον δεν θα ξαναγοράσει από το διαδίκτυο και αυτό φυσικά έχει αρνητικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή οικονομία. Στο παρελθόν ε, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ αυτές οι διαδικασίες, αλλά τώρα χάρη στο νέο σύστημα θα αλλάξει αυτό. Επομένως είμαι υπέρ αυτής της νέας νομοθεσίας. Το 82% των καταναλωτών παρόλα αυτά δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο για τις μικροδιαφορές. Παραδείγματο ε, χάρη όταν ε, έχει υπάρξει ζημία. Νομίζω όμως ότι αυτή η νομοθεσία θα βοηθήσει την κατανάλωση. Κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Ρίμπλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όλοι θέλουμε η Ευρωπαϊκή, να υπάρξει η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί εδώ και χρόνια να παραμερίσει όλα τα εμπόδια. Όλοι θέλουμε επίση να αξιοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό της ψηφιοποίηση για τους ε, πολίτες, για τις επιχειρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό λοιπόν συγκαταλέγονται και οι υπηρεσίε ε, και τα προϊόντα να μπορούν να παρέχονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό τι σημαίνει ότι όταν υπάρχουν και διαφορές θα πρέπει να μπορεί να υπάρχει και ένας απλός τρόπος εκδίκαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτόν ακριβώς το στόχο προσπαθεί να πετύχει το έγγραφο το οποίο θα ψηφίσουμε αύριο. 25 χρόνια περίπου μετά από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ενέας Αγοράς, το 2007 εισήχθη ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ε, έχουν ένα σύστημα λοιπόν επίλυσης τέτοιων διαφορών. Αυτό που τώρα θέλουμε να πετύχουμε και διαπραγματευτήκαμε χάρη στην εισηγήτρια και στους εισηγητές όλων των ομάδων ε, αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν ε, λοιπόν ε, πολύ γλώσσα έντυπα, μπορεί κανείς να ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή της προσφυγής ηλεκτρονικά και θα πρέπει και τα τέλη να είναι ανάλογα. Αυτό που σημαντικό είναι το ανώτατο όριο σε ό,τι αφορά την ε, ορισμό των μικροδιαφορών να είναι στα 5.000 ευρώ και στα 10.000 ευρώ όπως προέβλεπε αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο ακούσαμε επίσης είναι ότι η διαδικασία δυστυχώς ακόμα δεν ε, εφαρμόζεται, δεν χρησιμοποιείται επαρκώς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προβάλλουμε στο κοινό αυτό το μέσο προκειμένου να αξιοποιήσουμε πλήρως την ενιαία αγορά και αυτό εναπόκειται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και σε εμά του ευρωβουλευτέ Θα το κάνουμε λοιπόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νεγκρέσκου είναι ο επόμενο. για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ και θα ήθελα καταρχά να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έγγραφο το οποίο μας παρουσίασε σήμερα. Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα αυτή η έκθεση για την απλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επίλυσης Μικροδιαφορών και της κατάρτισης ενός κοινού συστήματος για την πληρωμή. Σε ό,τι αφορά τη μείωση στα 5.000 ευρώ, θεωρούμε ότι θα ευνοήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τώρα ε, διστάζουν σε πολλές περιπτώσεις να ε, προσφύγουν γιατί το τρέχον όριο του 2.000 ευρώ καλύπτει ένα 20% των περιπτώσεων, ενώ ότι η αύξηση σε 5.000 ευρώ θα αυξήσει το ποσοστό σε 40% αυτό. Και έτσι λοιπόν θα αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητες της νέας αγοράς. Ε, υποστηρίζω επίσης πλήρως την ιδέα να αξιοποιηθούν πλήρως τα ηλεκτρονικά συστήματα για να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή διαδικασία. Είτε μη πρόκειται για την υποβολή της προσφυγής, είτε πρόκειται για την διαδικασία εκδίκαση. Οι νέε τεχνολογίε συμβάλλουν στην μεγαλύτερη διαφάνεια και στην καλύτερη πρόσβαση στου ευρωπαϊκού μηχανισμού. Επίση, άλλα τρία στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκθεση. Σημαντικά, θέλω να το υπογραμμίσω. Μείωση των δικαστικών τελών ε, ε δωρεάν ε, αρρωγής και επίσης ε, σε ό,τι αφορά το δικαστικό φόρο να ε, υπάρξει καλύτερη προσαρμογή. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Δύο λεπτά. Η κυρία Κομοντίνη Κακία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς βλέπουμε μέσω αυτού του κανονισμού μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των απλών ανθρώπων αλλά και των επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν δυσκολίες προσφυγής λένε ότι οι δικαστικές διαδικασίες δεν είναι αποτελεσματικές και είναι και πάρα πολύ δαπανηρές. Αυτός ο κανονισμός προσπαθεί να τα εμπόδια τα οποία εμποδίζουν τους Ευρωπαίους πολίτες να βρουν λύσεις στις διασυνοριακές τους διαφορές. Προσπαθεί να ρυθμίσει το κόστος αλλά και να διευκολύνει την πρόσβαση στη δικαιοσία μειώνοντας την γραφειοκρατία με μια πιο απλή και πιο ταχεία διαδικασία. Πρόκειται για μια διαδικασία fast track, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν πλήττει και δεν μειώνει την δικαιοσύνη. Βελτιώνονται οι διαδικαστικές πτυχές, αυξάνεται η ταχύτητα και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα για τις ε, συναλλαγές στο διαδίκτυο, εκεί που δεν είναι πολλές φορές σαφής οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες. Είναι μια ταχεία διαδικασία επίλυσης αυτών των διαφορών, γι' αυτό και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να βαλτιστοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν στους πολίτες, απλοποιώντας την πρόσβαση και μειώνοντας το γραφειοκρατικό άχθος. Την ίδια ώρα βελτιώνεται η κατάσταση και των επιχειρηματιών αυτών, των εμπόρων, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες ε, των ψηφιακών συναλλαγών. Είναι πολύ σημαντικό για όλους αυτούς να εποφεληθούν από την εσωτερική ψηφιακή αγορά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν την διαδικασία Catch the Eye, δίνω το λόγο στον ε, κύριο Μπράντιν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτρο, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και όλους τους κοιόδης εισηγητές. Σας ευχαριστούμε για την εργασία σας για την εκθέση αυτή. Πιστεύω ότι η απλουστευμένη διαδικασία για τις μικροδιαφορές είναι ένα βήμα προς τα μπρος, προς την εισαγωγή κοινών κανόνων στις δικαστικές διαδικασίες στην Ευρώπη. Το ανώτατο όριο τώρα είναι 5.000 ευρώ και αυτό συντεριάζει με την οικονομική πραγματικότητα. Νομίζω ότι αυτό θα μας οδηγήσει σε καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού και τώρα αρκετοί πολίτες αλλά και μικρές και μεσές επιχειρήσεις ε, θα δράξουν αυτή την ευκαιρία. Και σε σχέση με τις μικροδιαφορές που σχετίζονται με το εργατικό δίκαιο. Αυτός ο κανονισμός θα παρέχει την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους να τους αποδοθεί δικαιοσύνη οπουδήποτε και αν ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται τώρα δηλαδή η δυνατότητα να πληρώσει κάποιος online και το να υπάρχει μία απλή γραπτή διαδικασία, όλες αυτέ είναι ευκαιρίε που θα είναι πάρα πολύ ελκυστικέ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομηθούν χρήματα και δεν θα υπάρξουν εμπόδια. Νομίζω ότι με αυτόν τον κανονισμό θα επιλύουμε με καλύτερο τρόπο τις μικροδιαφορές. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί ευρώ στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση που συζητούμε σήμερα είναι πολύ σημαντική καθώς εξετάζει τη θέσπιση διαδικασίας Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής όσον αφορά τις μικροδιαφορές συμφωνώ λοιπόν πως πρέπει να απλουστευτεί η διαδικασία διαταγής πληρωμής για τις μικροδιαφορές γιατί με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί το διασυνοριακό εμπόριο και οι συναλλαγές. επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ στη διαδικασία κατασχέσεων μισθών και συντάξεων που έχει επιβάλει η τρόικα με το μνημόνιο τρία στην ελλάδα. το ακατάσχετο μειώθηκε από τα 1.500 ευρώ στα 1.000 ευρώ με αποτέλεσμα το κράτος και οι τράπεζες να βάζουν χέρι στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φτωχοποιημένων ελλήνων επομένως στην ελλάδα η διαδικασία εκτέλεσης διαταγών πληρωμής μπαίνει ουσιαστικά στην υπηρεσία του μνημονιακού κράτους και των τοκογλύφων δανειστών. κυρία πρόεδρε από το βήμα της ευρωβουλής θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά πως οι αντιμνημονιακοί πολίτες θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την κατάργηση των μνημονίων στην ελλάδα τη διαγραφή του επονίδη του χρέους και την έξωση της τρόικας από την πατρίδα μας. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκίκορ για ένα λεπτό επίσης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κανονισμός αυτός έρχεται στη σωστή χρονική στιγμή και επιτρέπει καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Οι πολίτες μας δεν είναι δυνατόν να αποστερούνται των δικαιωμάτων τους. Και γι' αυτό λοιπόν αυτό αποτελεί ένα σωστό βήμα προς την ε, κατεύθυνση την οποία επιθυμούμε. το κόστος θα πρέπει να είναι ανάλογο με την αποζημίωση που επιδιώκεται και επίσης τα δικαστικά τέλη θα πρέπει να είναι και αυτά αναλογικά προς ε, το ποσό αποζημίωσης και φυσικά θα πρέπει να διακυβεύονται τα δικαιώματα του πολίτη. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου για παράδειγμα ο εργαζόμενος, ε, ο εργοδότης δεν, ε, τους μισθούς τα, και τις κοινωνικές παροχές στους εργαζομένους και φυσικά υπάρχουν πολλές διαφορές που προκύπτουν από διαδικτυακό εμπόριο και θα πρέπει λοιπόν οι πολίτες να διεκδικούν τα δικαιώματά τους που προκύπτουν από αυτές τις υποθέσεις. Ευχαριστώ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επίτροπο Γιούροβα. Για μια φορά ακόμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ, οι συμβιβασμοί που πετύχατε με το Συμβούλιο θα σημαίνουν ε, σημαντικά, νέα σημαντικά Οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν πιο συχνά τη διαδικασία επίλυσης μικροδιαφορών με χαμηλότερο κόστος και με μικρότερη διάρκεια για την εκδίκαση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας και μετά τη σημερινή συζήτηση είμαι αισιόδοξη ότι θα υπερψηφίσετε το συμβιβασμό που πετύχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Και τώρα το λόγο έχει η εισηγήτρια, η κυρία Γκέριγεντ Ούντεμπεργκ. E, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους για τα ευγενικά τους ε, λόγια απέναντι στη δουλειά μου. Πιστεύω ότι αυτό το νομοθέτημα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε ταχείες και μη δαπανηρές διαδικασίες. Μέχρι τώρα οι διαδικασίες δεν ήταν αποτελεσματικές. Πράγματι οι πολίτες δεν γνώριζαν αυτή τη διαδικασία. Ήταν μια διαδικασία πολύ ακριβή και πολύ συχνά οι πολίτες θεωρούσαν ότι λόγω της αθότητάς τους έπρεπε να πληρώσουν. Αντίθετα, με αυτή την ε, νέα νομοθεσία αντικαθιστούμε το παλιό νομοθέτημα. Η Επιτροπή Νομικών Θυμάτων ε, ομόφωνα ενέκρινε την έκθεση και θα ευχόμουν το ίδιο να συμβεί και αύριο στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Την εισηγητή ολοκληρώσαμε.